Hello everyone. Good afternoon. Um, I invite you to Ας αρχίσουμε τη συνάντησή μας, τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν θα ήθελα οι διερμηνείς να μας ε, διαβάσουν το μήνυμά τους, αλλά σας παρακαλώ πολύ να βάλετε τα ακουστικά σας. από την ε, ερμηνεία θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι βρισκόμαστε στην 35η ημέρα των διαπραγματεύσεων με την διοίκηση. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Ελπίζουμε να υπάρξει κάποια ανταπόκριση. αλλά προς το παρόν ε, ως κινητοποίηση δεν θα δώσουμε υπερβάση του προαθροισμένου ωραρίου. Και συνεχίζει η Πρόεδρος. Να... Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Εν όψη του μεγάλου φόρτου εργασίας οι συντονιστές θα προβάλλουν άλλες προθεσμίες για τροπολογίες, αλλά δεν θα υπάρξει προσχέδιο γνωμοδότησης και οι τροπολογίες θα συνταχθούν μαζί σε μια γνωμοδότηση εξ της Προεδρίας δηλαδή το πρόγραμμα ε, δορυφορικής ε, ε, σύνδεσης 25 Σεπτεμβρίου για την ΕΜΒΗ, ο μηχανισμός για την επίλυση νομικών διαφορών, ίδια προθεσμία 25 Σεπτεμβρίου 2018, το μέσο για την προενταξιακή βοήθεια και πάλι 25 ε, Σεπτεμβρίου στις 11. Επίσης η σήμανση των ελαστικών 25 Σεπτεμβρίου στις 11 και προαπαιτήσεις για την ε, έγκριση οχημάτων και αυτοκινούμενων οχημάτων καθώς και των ρημουλκών τους και των συναφών ε, συστημάτων μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας 26 Σεπτεμβρίου του 2018 και ως προς την, ε, το μέσο γειτονίας ανάπτυξης και διεθνής, διεθνούς συνεργασίας 26 Σεπτεμβρίου στις 11. Και πάλι, επειδή υπάρχει πολύ, μεγάλη, με πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, προβλέπεται έκτακτη συνάντηση στο Στρασβουρό την 1η Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 9 για να ψηφίσουμε ορισμένες επίγουσες γνωμοδοτήσεις. Θα σας δοθεί εν ευθέτω χρόνο η ημερήσια διάταξη. Επίσης υπάρχει και η έκθεση της επίσκεψης της ΕΜΒΗ στη DG Sante ε, στο Δουβλίνο και στο Grange της Ιρλανδίας που έγινε από τις 4 έως τις 6 Απριλίου. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες και φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την συνεδρίαση μέσω web streaming. Επίσης έχουν ε, διανεμηθεί οι γνωμοδοτήσεις και συστάσεις των ε, συντονιστών, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Πρώτο θέμα, λοιπόν, είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Όλα τα τμήματα. Θα πω και εγώ λίγα λόγια, στις 23 Μαΐου η Επιτροπή πρότεινε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2019, τον έκτο προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια του πολιετούς 14-20 που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την ασφάλεια. Μιλάμε για 166 δις στις υποχρεώσεις, δηλαδή συν 3% σε σχέση με το 2018 και 149 δις στις πληρωμές, δηλαδή και πάλι ε, ένα 3% επιπλέον. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια για να φτάσουμε στο στόχο του 20% για ε, τα κονδύλια που σχετίζονται με το κλίμα, δηλαδή 21% των συνολικών ε, υποχρεώσεων μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού 2019 που σχετίζονται με τα κλιματικά. Μιλάμε για 19,3% ε, ε, συνολικά και επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε την ε, βιοδιαφορετικότητα και στα πλαίσια των οργανισμών και του ε, ΡΙΜΙΤ θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια σε αυτούς τους οργανισμούς, έτσι ώστε να έχουμε μία προσέγγιση υπέρ της επιστήμης στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Επίσης, τα πιλωτικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα, έχουν, θα πρέπει να έχουν επαρκή χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του κύκλου ζωής. Έχουμε 33 ε, προτάσεις πιλωτικές και προπαρασκευαστικές δράσεις για ε, προαποτίμηση κατά τα τέλη του Απριλίου. Το Κοινοβούλιο έστειλε 344 προτάσεις. Στις 2 Ιουλίου ε, λάβαμε απάντηση από την Επιτροπή και στις προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα, αυτά τα προγράμματα θα αποτελέσουν μέρος του προϋπολογισμού 2019 και γι' αυτό θα πρέπει να υποβληθούν ως τροπολογίες επί του προϋπολογισμού μέχρι τις 11 Ιουλίου στις 11. Όπως και πέρσι η θέση του Συμβουλίου θα ε, ληφθεί πολύ αργά, δηλαδή την ίδια ημέρα με την προθεσμία στην ΕΜΒΗ και γι' αυτό θα υποβάλω τροπολογίες, δημοσιονομικές τροπολογίες για να αποκαταστήσουμε τον ε, προπολισμό του 2019 μέσα στα πλαίσια της εντολής της ΕΜΒ στις προτινόμενες ε, περικοπές του Συμβουλίου. Θα ήθελα τώρα να λάβετε το λόγο. Ο κύριος Πότς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση γιατί θα πρέπει σε μια άλλη επιτροπή να παρουσιάσει τις θέσεις της. Ευχαριστεί την εισηγήτρια την κυρία Βαλεάν και θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα όριο και στα πλαίσια της ΕΜΒΗ θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτές τις τροπολογίες. Μιλάμε για ε, σωστή χρηματοδότηση του 2000 ε, στον προϋπολογισμό του 2019 και θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα ενσωματώσουμε αυτή την πολιτική στις άλλες. Η Natura 2000 θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις συνέργειες χρηματοδότησης. Ως προς τον προϋπολογισμό ε, του 2019 δεν θα πρέπει να στάθουμε στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ξεχωριστό μέσα στα πλαίσια του πολιετούς. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε προς τον κύριο Βιώτη ότι έχει μεγάλη σημασία να το θεωρήσουμε αυτό το έργο ως πρόκριμα έτσι ώστε να υπάρξει η επαρκής χρηματοδότηση για να προωθήσουμε την πολιτική υγείας και ασφάλειας σε σχέση με τους οργανισμούς και τον αυξανόμενο προϋπολογισμό τους, η κυρία Κάντενμπαχ μαζί με την κυρία Βαλεάν θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι ε, ε, πόροι και ιδιαίτερα αυτό αφορά το κεφάλαιο των ανθρώπινων πόρων και θα υποβάλει τροπολογίες. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Κάντενμπαχ σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων για τους οργανισμούς μέσα στα πλαίσια του μεταναστευτικού και του έλεγχου των συνόρων. Θα πρέπει να συνδράμουμε με την ΕΦΣΑ, η οποία θα πρέπει να συνδράμει για να δούμε ποιες είναι αλλαγές, οι αλλαγές στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Ο κ. Ομαρτζή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των ε, μελημάτων μας ε, σε αυτή την Επιτροπή. Και αυτό αφορά και την ομάδα μου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των εγγραφών στον προϋπολογισμό και την ε, δινή κατάσταση στον τομέα της οικολογίας και ιδιαίτερα της βιοπικιλότητας. Για αυτούς που μας ακούν στο διαδίκτυο θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Το 100% των ζωικών ειδών ε, εξαμφανίζονται ημερησίως και το 41% των αμφιβίων και το 40% των θηλαστικών θα μπορούσαν να εξαφανιστούν. Επίσης, οι κοραλιογενείς νήσοι έχουν έχουν συρρυκνωθεί και 77% των 60% ε, συγγνώμη, συγγνώμη των ε, ε, ηχθείων έχουν ε, μειωθεί, έχουν εξαλειφθεί μέσα στα πλαίσια των 40 ε, τελευταίων ετών. Υπάρχει ένας κόκκινος ε, κατάλογος των ε, Ηνωμένων Εθνών που έχει επικαιροποιηθεί το 2016. Θεωρούνται ήδη υπό απειλή. Και 5.583 ήδη απειλούνται με εξαφάνιση και 11.000 θα εξαφανιστούν εντελώς. Αυτό αφορά και τους ελέφαντες της Αφρικής που δυστυχώς έχουν μειωθεί κατά 50% τα, τις τρεις τελευταίες ε, γενιές. Στη Γαλλία, από όπου προέρχομαι, έχουμε μία ηλικιώδη μείωση των ε, οδικών πτηνών 60% τα τελευταία 10 χρόνια και επίσης ε, ένα μεγάλο ποσοστό κοριδαλών έχουν ε, εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Εάν λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία, το 2050 δεν θα υπάρχει ούτε ένα ψάρι, ούτε ένα μαλακόστρακο, ούτε τίποτα για την επίσημη αλία. Πρόκειται για μία ε, αδυσόπιτη κατάσταση για την ανθρωπότητα και γι' αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις που να είναι στο ύψος των περιστάσεων από δημοσιονομικής πλευράς. Όταν δείτε το ε, εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το LIFE, για την προστασία της βιοπικιλότητας, βλέπετε ότι για το 2019 αποτελεί το 0,3% του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι με βάση αυτό το πανόραμα βλέπετε πως οι απαντήσεις του προϋπολογισμού είναι ανεπαρκείς. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένα ποιοτικό άλμα, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το διακύβευμα που αφορά την επιβίωση της βιοπικιλότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν Θέλει κανένα συνάδελφο να πάρει το λόγο. Αν όχι, να ακούσουμε τους εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταρχάς έχουμε την κυρία Κοτουκάουτσκα. από τη Γενική Διεύθυνση ΕΒΗ. Thank you very much uh, for giving me σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και σημείωσα όλες τις ανησυχίες σε ό,τι αφορά την διαπικιλότητα και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος ακόμη και για τα σημαντικά αυτά στοιχεία. Θα δώσω γραφτές λοιπόν απαντήσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Το πρόγραμμα Live για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει δρομολογηθεί απόλυτα. Έχουν ε, υπογραφεί τα πρώτα προγράμματα για το 2014 και 2015. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης υλοποίηση και δεν έχουν ε, φανεί ακόμα 100% τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε από την, κυρία, από την Γενική Διευθυνσή Σάντα, ο κύριος Ντερκλέρκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Συμφωνούμε με το σχέδιο γνωμοδότηως. να πούμε ότι κάθε εξωτερική υπηρεσία κάθε χρόνο υποβάλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο πρόγραμμα που τονίζει τις προτεραιότητες της υπηρεσίας για τα επόμενα χρόνια. Και εξ όσων γνωρίζουμε, το προσωπικό που διαθέτει κάθε υπηρεσία συνάδει με τις αρμοδιότητες. Μάλιστα, και τώρα ο κ. Φανχόλεμπικ από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Σας ευχαριστώ πολύ από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Action. Να πω δύο λόγια για το θέμα της ε, οριζόντιας και εγκάρσιας εφαρμογής του θέματος του κλίματος. Ήταν μια πρωτοποριακή, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα σε ό,τι αφορά την ένταξη του θέματος του κλίματος ε, αυτό που το πω. Ήταν φιλόδοξο στόχο, συμφωνούμε, αλλά νομίζουμε ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έγινε καλή δουλειά και ότι αυτό μα βοηθάει. Να περάσουμε στην ε, οικονομία χαμηλής, ε, χαμηλού άνθρακα που θέλουμε να έχουμε πετύχει μέχρι το 2050 σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό εξ αρχής, ε, όχι μόνο των οικονομικών προγραμμάτων της Ένωσης, αλλά και των πολιτικών της Ένωσης. Και πιστεύουμε ότι αυτή η πρόβλεψη το 19,3% στον τρέχον πουδουπού, σημαίνει ότι στο εγχείρημα αυτό θα έρθει και με επιτυχία. Και ενδεχομένω να μπορούμε να πετύχουμε κιόλα, γιατί έχουμε ακόμα και ένα έτο που υπολείπεται το 2020, μέχρι το 2020. Άρα μπορεί ακόμα να πετύχουμε τον στόχο του 20% που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και για την υποστήριξή σας υποβολή τραπολογιών μέχρι και για την γραμματοδότηση και για την προπολογισμό η 11η Ιουλίου. 11 το μεσημέρι, το πρωί. Και θα ψηφίσουμε 30 Αυγούστου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και έτσι ολοκληρώθηκε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα Έκθεση της κυρίας Καμπεσόν Ρουής, την οποία όμως δεν τη βλέπω. Να περιμένουμε κάνα δύο λεπτάκια. I'm told that Θα καταφτάσει σύντομα, με ενημερώνουν. Δεν μπορούμε δυστυχώς να αρχίσουμε χωρίς αυτήν. Uh, λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βλέπουμε τις ε, τροπολογίες για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011-2024. Η συγγήτρια είναι η κυρία Καμπεθόν Ρουή. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, señora Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω... Έχουμε 529 τροπολογίες συνολικά και η γενική αξιολόγηση είναι ότι έχουν αλλάξει ορισμένες θέσεις δραστικά που θα σχολιάσω, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές ουσίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συνένεση. Θα ήθελα να σταθώ στις ε, πτυχές που οδήγησαν σε μεγαλύτερες δυσκολίες. σε σχέση με την εισαγωγή των ιατρικών μηχανημάτων κατά υποχρεωτικό τρόπο καθώς και τον αποκλεισμό σε εθελούσια βάση, κάναμε μία πρόταση συμβιβασμού, την οποία θα αξιολογήσουμε, γιατί θεώρησα ότι θα έπρεπε να εργαστούμε επί του θέματος αυτού σε σχέση και με την ε, φιλόδοξη ε, θέση της Επιτροπής. Όταν μιλάμε για medical devices θα πρέπει να έχουμε ενιαία μεθοδολογία. Το ένα άλλο ουσιώδες ζήτημα είναι πώς θα εγκριθούν οι συμφωνίες με βάση την αξιολόγηση. Εγώ μιλούσα για δύο τρίτα όταν υπάρχει συνένεση ή με ειδική πλειοψηφία εκεί που χρειάζεται. Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία που θα μπορούσαν να γύρουν δυσκολίες αλλά δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε σε μία συμφωνία καταρχήν. Επίσης, το άρθρο 8 που μιλάει για την εθελούσια υποχρεωτική βάση ή αξιολόγηση από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά κατά πλειοψηφία Θέλουμε να κρατήσουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα και τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για αυτές τις αξιολογήσεις. Δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα ως προς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα για να συμπλέψουμε ενδεχομένως και με το Συμβούλιο, αλλά στόχος ε, της πρότασης είναι να εναρμονίσουμε τα κλινικά και επιστημονικά κριτήρια και στον ε, ε, κλινικό τομέα δεν θα μπορούσαμε να παρέμβουμε γιατί υπάρχει επικουρικότητα. Μετά το άρθρο 22 αφορά τη μεθοδολογία που αφορά το, τα κλινικά δεδομένα και τα επιστημονικά για να υπάρχει η κατάλληλη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και ε, δεν υπάρχουν υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους εθνικούς ε, οργανισμούς, έτσι ώστε σε σχέση με τις κατεκτέλεση ε, πράξεις να μπορέσει και η Κομισιόν να δράσει με βάση τους οργανισμούς αξιολόγησης. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα δράσουν μέσω του εθνικού οργανισμού για να υπάρχει εμπιστοσύνη και για να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, δεν υπάρχει καμία ε, ομάδα, πολιτική ομάδα που αντιτίθεται σε αυτή την ε, πρόταση. Επίσης θα πρέπει να, να δούμε πώς θα επιλέξουμε αυτά τα ιατρικά μηχανήματα και αν θα ακολουθήσουμε την απλή πλειοψηφία, την πλειοψηφία δύο τρίτων ή την ειδική. Ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων, όμως ε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ των ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης ηγητές, η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Ε, merci Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία Καπιθόν Ρουή, η οποία είναι η συγκεκριά μα και έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Και να την ευχαριστήσω κυρίω για την ε, συνεργασία και το πνεύμα συνεργασία με το οποίο εργάστηκε. Μα. εξήγησε λοιπόν τι έγινε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα πιο απαραίτητα σε ό,τι αφορά καταρχά τη στρατηγική. Ξέρουμε ότι σε μεγάλο κομμάτι των κρατών μελών στο Συμβούλιο υπάρχει διάθεση συνεργασία δεν θέλουν ε, υποχρεωτική εισαγωγή των συστημάτων ε, στην τεχνολογία υγείας. Καταλαβαίνουμε φυσικά ε, τις ανησυχίες τους και το, την ανησυχία για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματο, αλλά να μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα έπρεπε απαραίτητο, αν θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, να διατηρήσουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινής αξιολόγησης να απαντήσουμε στο σωστή ανησυχίε που εκφράστηκαν σε ό,τι αφορά την ομάδα συντονισμού προκειμένου να υπάρχει πραγματική συνεργασία και να έχουν πραγματικά τα κράτη-μέλη τον έλεγχο. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορες τροπολογίες. Να. Να διευκρινίσουμε του κανόνες του άρθρου 8 για να δώσουμε πιο πολύ ευελιξία και για να διευκρινίσουμε τι είδους ε, συνεργασία συμπληρωματική μπορεί να υπάρξει για να αποφευθεί οποιαδήποτε νομική αβεβαιότητα. και τα άλλα, πιστεύω όπως και άλλοι ότι η μεθοδολογία αξιολόγησης ε, στο άρθρο 22 θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Είμαι αντίθετη. Ωστόσο, στο να είμαστε υπερβολικά ε, διευκρινιστικοί και περιοριστικοί για να μην επιτρέψουμε τελικά να υπάρχει προσαρμογή της μεθοδολογίας ανάλογα και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Επιμείνουμε επίσης στην ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια και προσβασιμότητα στα δεδομένα. Κατανοώ φυσικά τις απαιτήσει αυτές, αλλά να υπάρχει και ένα διστάθισμα, μια ισορροπία σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει και η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε ό,τι αφορά τα προσωπικά των τα οποία είναι εμπορικώ αξιοποιήσιμα, σε έναν ε, τομέα πολύ ανταγωνιστικό είναι γεγονό ε, κατά τη διάρκεια των, των ε, διαβουλεύσεων και στην εμπορική φάση. Τέλο, να αναφέρω δύο περιπτώσει. Το θέμα των διατάξεων των ιατρικών διατάξεων και των φαρμάκων σε ό,τι αφορά τα φαρμακά θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει κοινή κλινική αξιολόγηση για να μην υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά τα φάρμακα τα οποία τα οποία δεν είναι κατοχυρωμένα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει αντιμετώπιση, αλλά να επιτρέπει και την διαφοροποίηση των υγειονομικών συστημάτων σε ό,τι αφορά και τη συμπληρωματικότητα των ε, μεθοδολογιών. Αυτό σε αθελούσια βάση. Ή, βάση, περιπτώσει, θα πρέπει να προβλέπετε παρέμβαση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, ε, την ε, συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια μέση λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια με την οποία η συζήτηση ήταν πραγματικά πολύ άνετη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πιέτσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας ε, παρουσίασε και το πεδίο εφαρμογή και το πώ έχει η κατάσταση και πώ πήγαν τα πράγματα στην Επιτροπή. Ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία δεν είναι ιδιαίτερω ε, θετικά στο να δεχτούν ε, αυτέ τι αλλαγέ και μιλούμε για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Αυτέ οι γνωμοδοτήσει έχουν παρουσιαστεί ξεκάθαρα, οπότε πρέπει να είμαστε κάπω ευέλικτοι και ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί σε άλλη περίπτωση μπορεί να καταλήξουμε σε ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα ή σε μια πολύ φιλόδοξη πρόταση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να την απορρίψει τελικώς. Οπότε το Συμβούλιο μπορεί να μην ακολουθήσει τη δική μας γραμμή ή μπορεί να εμπλακεί στους, στα γραφειοκρατικά γρανάζια του Συμβουλίου όλη αυτή η προσπάθεια. Συμφωνώ ότι το HTA είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τεράστια πρόκληση και ξέρουμε ότι υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη υπηρεσίες και μάλιστα σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν και πάνω από μία υπηρεσίες. Μπορεί να είναι εθνικά ιδρύματα, μπορεί να είναι εμπορικά ιδρύματα και έχουν την, ε, το δικαίωμα να μπορούν να αξιολογούν την ιατρική τεχνολογία. Οπότε να κάνω δύο σχολεία προς αυτό. Καταρχάς αυτό είναι ε, υποχρεωτικό και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτός ο υποχρεωτικός χαρακτήρας είναι άτεγκτη προσέγγιση κυρίως όταν ε, πρόκειται για την ε, τεχνολογία υγείας και την πρόληψη, τη διάγνωση κτλ. Εδώ νομίζω ότι θα χρειαζόταν κάποιο είδου αξιολόγηση ή κάποιο είδου υπολογισμό για την ε, τεχνολογία υγεία στα κράτη-μέλη. Βεβαίω, ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι και ανεξάρτητα όταν ε, πρόκειται για την διαχείριση του ιατρικού, του ε, ιατρικού τομέα, την χρηματοδότηση κτλ. Υπάρχουν συμμετοχές ε, των ε, ιατρών, των ασθενών, των ε, ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο υποχρεωτικός χαρακτήρας θα αποτελέσει το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της πρότασης. Και δεν νομίζω ότι αυτά τα πρότυπα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Και δεύτερον, οι ιατρικές συσκευές. Έχουμε ε, χιλιάδες, ε, χιλιάδες συσκευές που μπορεί να είναι πολύ μικρές, που μπορεί να μην είναι πολύ περίπλοκες στη χρήση τους ή τη λειτουργία τους, που δεν προσθέτουν κατά ανάγκη τόσα πολλά στην ιατρική τεχνολογία, μπορεί να κάνουν κάτι πάρα πολύ βασικό. Ας πούμε, έχουμε ιατρικές συσκευές οι οποίες ε, ε, εκλείουν ενέργεια για κάποιες, ε, ή ραδιενέργεια για κάποιες σοβαρές ασθένειες ή ας πούμε για καρκινικούς όγκους. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά και απ' την άλλη είναι σαφές ότι η αξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας είναι τόσο ταχεία που ακόμη και αν βρούμε μια πολύ καλή μεθοδολογία για να την ρυθμίσουμε σε κάποιες υπηρεσίες από κοινού και με την συντονιστική ομάδα πάντα θα υπάρχει μία περίπτωση όπου η ε, τεχνολογία θα είναι ένα βήμα μπροστά από μας. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν μετά τα ε, Ινστιτούτα των Κρατών Μελών να δουλέψουν πάνω στο κάθε επιμέρους πρόβλημα. Και ας είμαστε προσεκτικοί. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέλουν ε, διαφάνεια. Πρέπει να δούμε πόση διαφάνεια και πόση εμπιστευτικότητα θα υπάρξει. Για να μην μιλήσω για τα φάρμακα, Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε και το ε, δίκαιο ε, για τα ε, διπλώματα Ε, Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Όλος ο καυγάς που γίνεται, κυρίω όταν πρόκειται για την δημιουργία νέων φαρμάκων, α πούμε, φάρμακα για τους καρκινικούς όγκους, ή για άλλες ε, ασθένειες, αυτά τα φάρμακα που σχετίζονται με την ε, μικροβιακή αντίσταση ε, κοστίζουν πολλά, πρέπει να υπόκεινται σε ένα πολύ μακροπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα για τα συγκεκριμένα τα δεδομένα φάρμακα ή την ιατρική συσκευή για να μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε. Οπότε το να βρούμε μια χρυσή τομή μάλλον θα είναι δύσκολο και μάλιστα εγώ είμαι και πολύ διστακτικός για το σύνολο της πρότασης. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές ε, λύσεις, θα έχουμε κάποιο περιθώριο ελιγμών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί να είναι αποδεκτό και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην είναι όσο φιλόδοξο θέλαμε να είναι στην αρχή, αλλά ελπίζω ότι τελικώ θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι αποδεκτό από το Συμβούλιο, γιατί τα κράτη-μέλη θα έχουν πολλά να πούνε σε αυτή την πρόταση. Και αν διαβάσετε και κάποιες ε, γνωμοδοτήσεις από διάφορες ε, αντιπροσωπείες του Συμβουλίου, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Αυτά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Κάναμε και μια σκιώδη συζήτηση, συνάντηση. Ήταν πολύ ωραία, ήταν λεπτομερέστατη η συζήτηση που κάναμε. Αυτό που δεν κάναμε είναι να σας πούμε τι συζητήσαμε για να μπορέσετε να το σχολιάσετε. Σήμερα την Πέμπτη θα ξανασυνδυθούμε ε, με τους κοιόδες, οπότε είναι πολύ εντατική η δουλειά μας γιατί το θέμα είναι πολύ απαιτητικό. Πολλοί μίλησαν, τα κράτη πολλά κράτη μέλη δεν το θέλουν καν την πρόταση αυτή. Ε, εμένα η ομάδα μου η πολιτική στο, από την Βουλή μου είπε ότι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν δεν το θέλουμε, ε, μην ξεκινήσετε καν διαπραγματεύσεις γιατί έχουμε και θέμα θέματα ε, υπά... αυτό το θέμα είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών από τη μια. Από την άλλη έχουμε στην Ευρώπη την ελεύθερη κινητικότητα εμποριών, εμπορευμάτων ανθρώπων και υπηρεσιών. Ε, και εδώ έχουμε ένα θέμα που περιλαμβάνει και τα τρία. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ενοποιήσουμε τα πράγματα όπου είναι σκόπιμο, αντί να έχουμε 27 ή 28 διαφορετικέ μεθόδου αναγνώριση κτλ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει η πρόταση αυτή. Αλλά για τους λόγους αυτούς πρέπει να πω ότι το άρθρο 8 πρέπει να είναι ευέλικτο για τα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι επιπισμένη ότι πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή την ε, πρόταση να την ε, ολοκληρώσουμε σε έναν ε, καλό τριμερή διάλογο, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να είναι διατεθειμένα να διαπραγματευτούν όταν μπορέσουμε να του δώσουμε και αυτόν μια, αλφα ευελιξία. Οπότε πρέπει να δούμε τι είναι τι, τι είναι υποχρεωτικό και τι θα είναι θελούσιο για τα φάρμακα σίγουρα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σύστημα, ε, θελούσιο για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ε, αυτό που είπε βεβαίως η κυρία ε, Γκροστέτ είναι σωστό. Τα φαρμακευτικά προϊόντα ήδη υπόκεινται σε συγκεκριμένο κανονισμό για την εφαρμογή από το 2020 και εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία για την κλινική αξιολόγηση κτλ. Τα οποία εδώ ουσιαστικά θα δημιουργούσαν διπλή δουλειά. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Το άλλο, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη κάνουν αυτό που κάνουν ήδη για τα φάρμακα. 1% είναι το ποσοστό αυτό. Και μετά τα κράτη είναι υπεύθυνα για, την, για τον καθορισμό των τιμών. Ο κανονισμός όμως αυτός δεν χρησιμοποιεί τόσο εργαλείο για να πετύχουν αυτή την ε, διάταξη. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει εθελούσιο στα, για τα κράτη-μέλη. Μετά, Σίγουρα αυτό το HTA δεν θα είναι αρκετά προικοδοτημένο. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό και αυτό που είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να περάσει από κάποια κρατημέλη. Για τα υπόλοιπα θεωρώ ότι πρέπει να είναι εθελοντική ανταλλαγή και όχι υποχρεωτική. Μετά κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι καλά. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορισμένος. Είναι ο συντονιστής, ας πούμε, της όλης προσπάθειας. Εγώ θεωρώ ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη προ αυτό. Είναι σημαντικό να εμπλέκονται και άλλοι ε, εμπειρογνώμονες εδώ και επίσης για την πλατφόρμα των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να τη συζητήσουμε, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Νομίζω ότι είναι λίγο ανισόρροπο έτσι όπως προτείνεται στην πρόταση. Είναι καλό να έχουμε και τις ε, μη κυβερνητικέ και τους εκπροσώπους των ασθενών κτλ. Αλλά η προστασία των καταναλωτών χρειάζεται να είναι παρούσα. Μπορούμε να το συζητήσουμε βεβαίω αν θέλετε. Και απ' την άλλη, οι εμπειρογνώμονε, πάντα για του εμπειρογνώμονε είναι σημαντικό να, και για του εκπροσώπου των παρασκευαστών να είναι ουδέτεροι, να μην έχουν δηλαδή δικά τους ε, ε, συμφέροντα τα οποία να θέλουν να ε, εξασφαλίσουν, αλλά τώρα να τους αποκλείσουμε και τελείως νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Ήδη είδαμε ότι στα φάρμακα μπορεί να είναι καλό να εμπλέκονται διάφορες φωνές που μπορεί να είναι από την έρευνα ή από τη βιομηχανία. Πρέπει να έχουμε την απαραίτητη πυρογνωμοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει ακόμα να το συζητήσουμε. Άλλα δύο σημεία. Διαφάνεια, το είπα πιο πριν. Γενικώ πάντα θεωρώ ότι είναι σημαντική η διαφάνεια και πρέπει να δούμε που θα, ε, τι θα γίνει με τα δεδομένα που δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Επίση τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τα προστατέψουμε, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και γενικώ θεωρώ ότι είναι αρκετά τεχνική η δουλειά που έχουμε, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική για του πολίτε τη Ευρώπη. Θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα βρούμε καλέ συμβαστικέ προτάσει. και για τα ε, ε, φαρμακευτικά προϊόντα, αν θα είναι υποχρεωτικό ή όχι, για το πεδίο εφαρμογή. Σίγουρα θα ε, καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Χαίρομαι λοιπόν για την περαιτέρω συνεργασία μα και όσο καλύτερα εκπροσωπήσουμε τις θέσεις μας, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι που να καλύπτει τους περισσότερους, αν όχι όλους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, συγκριτή και του Σκιώδη ε, και την κυρία Γκροστέτ ε, από το ΕΛΚΑ. Θα ήθελα να υποστηρίξω πολλά από αυτά που ακούσαμε πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και να κάνω και κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις σε ό,τι αφορά τα πιο αμφιλεγόμενα και ακαθόδη ζητήματα. Επί της αρχής λοιπόν. Όντως, είναι σημαντική η πρόταση. Εγώ και εγώ φυσικά στη Γερμανία βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τους εθνικούς βουλευτές και συχνά βλέπουμε ότι και στη Γερμανία και σε άλλα κρατημέλη υπάρχει έντονη αντίσταση και αυτό επικεντρώνεται σε κάποια περιορισμένα σημεία. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή η αντίδραση σε όλη την πρόταση. Α, θέλουμε να δούμε πώς θα κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις για τα καθόδη ζητήματα. Όντως θα πρέπει να αποφευθεί η διπλή δουλειά, η αλληλεποκάλυψη καθηκόντων. Να υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οργάνωση. Το άρθρο 12 και 6. διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φάρμακων και του HDA. Αν γίνει σωστά, θεωρώ ότι θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα την ε, βιομηχανία και θα επικεντρωθεί πραγματικά η βιομηχανία σε ωφέλιμα προϊόντα που βοηθούν τον ε, ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν ε, αξίζει τον κόπο και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο διάλογο αυτό με πολλού συναδέλφου. Ε, καταθέσαμε από κοινού κάποιε τροπολογίε. Το πρώτο, η πρώτη ομάδα τροπολογισμών για το opt-out. Ε, εθελούσια ή υποχρεωτική φύση. Εγώ θεωρώ ότι καταρχά θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για να μην υπάρχει τέτοια τέτοιο διχασμό. Για κάποιον που παράγει ένα προϊόν, ε, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να προβλέψουμε. Να υπάρχει και ευρωπαϊκή διαδικασία και 27 διαφορετικέ εθνικές διαδικασίε. Να είναι λοιπόν καταρχάς να υπάρχει opt-in. Να υπάρχει δυνατότητα όμως opt-out αν δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν οι εθνικέ διαδικασίε, ε, θεραπευτικές διαδικασίες στην ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή δυνατότητα σε περίπτωση που υπάρχουν πέντε διαφορετικέ διαδικασίε ε, να υπάρχει δυνατότητα να αντιτριθουν opt Opt-out δηλαδή. Ενίσχυση λοιπόν του, opt-out σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι όπω θέλει καθένα. Πώ θα αποφασίζει η ομάδα συντονισμού τώρα. Μία συζήτηση. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει με πλειοψηφία, απλή πλειοψηφία. Η κυρία Καμπεσόν ζητήσε ε, πλειοψηφία δύο τρίτων. Δεν έχει νόημα θεωρώ αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει ένας απλός ε, κανόνας ε, στις συνθήκες. Η ειδική πλειοψηφία. Πολύ απλά αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Είναι κάπου ανάμεσα στην απλή πλειοψηφία και στην πλειοψηφία δύο τρίτων. Για αυτά που αναφέρεται δεν θα μιλήσω άλλο. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι πολύ φιλοδόξη και στοχευμένη γιατί επιμένει στην διαδικασία εποπτείας και στον κανονισμό για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτά είναι δύο διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε τη διαδικασία για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Εδώ χρειαζόμαστε επιπρόσθετη ασφάλεια, αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Να μπορεί κανεί να εξετάσει αν πραγματικά υπάρχει ασφάλεια. Εδώ όμω δεν μιλάμε για ασφάλεια. Μιλάμε για την ε, ωφέλεια που έχει ένα προϊόν για τον ασθενή. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχει ένα επικίνδυνο προϊόν με παρενέργειες, για παράδειγμα, όταν ε, γίνεται εμφύτευση στον ασθενή. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διαδικασία παρακολούθησης. Να μην υπάρχει όμως αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα ή να μην συνεπάγεται πολύ κόστος. Από την άλλη μπορεί να υπάρχει κάποιο προϊόν όπου το θέμα της ασφάλειας δεν τίθεται καν. Εν τούτης μπορεί να υπάρχει υψηλό κόστος. Και θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε κατά πόσον δικαιολογείται αυτό το υψηλό κόστος και κατά πόσον υπάρχει όντω αντίστοιχη ωφέλεια για τον ασθενή. Άρα αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα συγχαίουμε. Θεωρώ ότι είναι παραπλανητική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό λοιπόν έκανα εγώ μια πρόταση ως εξή. Τα φαρμακευτικά προϊόντα καταρχά να εξαιρεθούν. Αναφέρθηκαν άλλωστε και τα επιχειρήματα. Είμαστε σε πρώιμη φάση και τα κρατημέλη δεν συμπεριλαμβάνουν στην ε, αξιολόγηση τιμή στο HTA, αλλά να συμπεριληφθούν τα θέματα αυτά όταν αρχίσει να γίνεται εθνική επεξεργασία των θεμάτων αυτών. Γιατί ο σκοπό μας είναι να αποφύγουμε έναν κατακαιρματισμό. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν HTA για τα εθνικά προϊόντα, δεν υπάρχει κατακαιρματισμό. Αν υπάρχει όμω ε, σιγά σιγά ξεχωριστή ε, διαδικασία ανακράτος, τότε θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Να το κοιτάξουν, ε, θεωρώ, οι συναδελφοί, το θέμα αυτό. Και είχα προτείνει από τη στιγμή που θα υιοθετήσουν πέντε κρατημέλη μια διαδικασία να θεωρηθεί ευρωπαϊκή. Αλλά είμαι ανοιχτό σε διαπραγματεύσει και συμβιβασμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισορροπημένη προσέγγιση όχι όλα έξω ή όλα μέσα και να υπάρχει μια αιτιολόγηση ανάλογα το προϊόν. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έκανα προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. If there is, uh, else... Ευχαριστώ. Άλλος κανείς που να θέλει το λόγο? Όχι. Η κυρία Αμπέλας από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Ευρωβουλευτή Καμπεθόν Ρουής για την ε, πολύ φιλόδοξη ε, έκθεση και για την δουλειά που έκανε και για τις απαντήσεις προς την πρόταση Κομισιόν. Είναι μια πρόταση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντά στο αίτημα που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, βασίζουμε την πρότασή μας σε έτη πολλά συνεργασίες που έχουν υπάρξει στα πλαίσια των διαφόρων κοινών δράσεων. Θέλω απλώ να μιλήσω για κάποια από τα θέματα που ακούστηκαν στη συζήτηση. Καταρχά το πεδίο εφαρμογή και το θέμα των ιατρικών συσκευών. Είδαμε ότι υπάρχουν αποκλίνουσε απόψεις στο Κοινοβούλιο για το αν θα συμπεριληφθούν ή όχι οι ιατρικές συσκευέ και ποια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Να αναφέρω εδώ ότι η Κομισιόν είχε κάνει μια ενδελεχή ε, διαβούλευση με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς πριν υιοθετήσει την πρόταση και άκουσε πάρα πολύ προσεκτικά στο, στη βιομηχανία παραγωγής οπότε, ε, ιατρικών συσκευών, οπότε θεωρούμε ότι έχουμε στην πρότασή μας καλύψει τις ανησυχίες που υπάρχουν από την βιομηχανία Επικεντρωνόμαστε δηλαδή σε περιορισμένο πεδίο για τις ιατρικές συσκευέ. Μιλούμε για αυτές που είναι υψηλού κινδύνου. Επιτρέπουμε μια ευελιξία σε ό,τι αφορά το χρονισμό της κοινή δουλειάς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μερίδιο της αγοράς είναι αυτό ακριβώς που είναι και έχουμε και μία προσέγγιση phase-in που, μπορούμε, που μας βοηθά να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες ε, ιατρικές συσκευέ για τα πρώτα χρόνια και μετά να διευρύνουμε το σύστημα αν θεωρήσουμε ότι είναι ε, καλά τα αποτελέσματα και είναι χρήσιμο. Επίσης θεωρούμε ότι οι ιατρικές συσκευέ θα πρέπει να, βρεθούν εντός του πεδίου εφαρμογή του, ε, του κανονισμού σύμφωνα και με τα όσα ακούσαμε από τη δημόσια διαβούλευση αλλά είναι πολύ, πιο, ε, πολύ, λιγότερη, ε, φιλόδοξη, πολύ λιγότερο φιλόδοξη αυτή η προσέγγιση από αυτή που έχουμε για τα φαρμακευτικά προϊόντα. οι ιατρικέ ε, διαδικασίε είναι πολύ πιο, οι εθνικές διαδικασίες για το HTA είναι πολύ πιο ανεπτυγμένε για τα φαρμακευτικά προϊόντα ε, σε σχέση με τι ιατρικέ συσκευέ. Γι' αυτό έχουμε περιορίσει το πεδίο εφαρμογή του άρθρο 5 για τι ιατρικέ συσκευέ, αλλά επιτρέπουμε και κάποια εθελοντική δουλειά να μπορεί να γίνει για τι ιατρικέ συσκευέ. Είτε είναι συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει για το άρθρο 19, είτε το εθελούσιο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Επίσης, να πω δύο λόγια για την, τον εθελοντικό ή τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρότασης. Νομίζω ότι το μήνυμα από την συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σε τεχνικό επίπεδο τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και να πω επίσης ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν προτείνει το άρθρο 8 και τα διάφορα στοιχεία που περιλαμβάνει η πρότασή της έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση των πόρων. Επενδύουμε στη δουλειά που κάνουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν κάνουμε λοιπόν αυτή την επένδυση θα πρέπει να αποφύγουμε επαναλήψεις όλων όσων έχουν ήδη γίνει από κοινού και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η κοινή αυτή δουλειά θα χρησιμοποιηθεί στα διάφορα κρατημέλη. Οπότε είναι θέμα βελτιστοποίησης των πόρων που έχουμε. Επίσης, ε, συμφωνώ με ε, αυτό που είπε η κυρία Γκροστέτ, ότι όντω όλα αυτά συνδέονται και στο να έχουμε μια διαδικασία από πλευρά κρατών μελών. Είναι συντονιστικός ρόλος, η εξασφάλιση ποιότητα τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Όλε αυτέ όλες αυτές οι πτυχέ θεωρώ ότι είναι επίση εξίσου σημαντικέ. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο δέσμευση από τα κράτη-μέλη, αλλά σεβόμενοι πάντα την εθνική αρμοδιότητα για τι αποζημιώσει, για την ε, τιμολόγηση κτλ. Μετά, και τη διαφάνεια. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι η διαφάνεια και η ανεξαρτησία είναι σημεία κλειδιά της πρότασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικές πτυχές. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι ίσως κάποια από τα δεδομένα μπορεί να είναι ιδιαίτερως ευαίσθητα, οπότε υπάρχει μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί κυρίως για τα δεδομένα, αλλά θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία πάντα με τους συγκεκριμένους περιορισμούς για τα δεδομένα. Και επίσης, ισορροπία μεταξύ του, του κατευθυντηρίου εγγράφου, του διατακτικού, του κοινωνισμού και των, των ε, εκτελεστικών πράξεων. Όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς θα συνδυαστούν. Έχουν υπάρξει κάποια στοιχεία στην πρόταση για τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, αλλά το θέμα είναι να εξεύρουμε την ισορροπία και να γνωρίζουμε και τα διάφορα νομικά καθεστώτα, εάν επιλέξουμε να μπει κάτι στα έγγραφα εργασία είτε, από, είτε στις, ε, στο διατακτικό του κειμένου είτε στην ε, καταξουδιώτηση ή την εκτελεστική πράξη. Και επίσης η συμμετοχή των κρατών μελών και των εθνικών δηλαδή εμπειρογνωμόνων ε, γίνεται και στην συντονιστική ομάδα και στην επιτροπολογία. που ούτως ή άλλως ε, υπάρχει λόγω του ότι θα υπάρξει εκτελεστική πράξη στο τέλος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η αλλως υπαρχει λογο του οτι θα Καβεσόν έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους σκιώδεις για την υποστήριξή τους. Θα ήθελα να πω ότι έχω δεχτεί πιέσεις ή σχόλια από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και καταλαβαίνω ότι τέτοιες αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν ε, δυσκολίες. Αλλά το Κοινοβούλιο, πέρα από αυτές τις ε, δυσκολίες που κατανοώ από ορισμένα κράτη-μέλη, διότι έχουν μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τα συστήματα υγείας και τις νέες τεχνολογίες, νομίζω ότι αυτή η πρόταση έχει μεγάλη σημασία για να παράξουμε περισσότερη Ευρώπη και να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις ε, τεχνολογίες υγείας. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτήν. Κατανοώ τις δυσκολίες ορισμένων κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τους ασθενείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν αυτή την πρόσβαση στις τεχνολογίες υγείας υψηλής ποιότητας. Νομίζω ότι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι αρκετά στεναρό. Όταν φτάσουμε στο τριμερή διάλογο, ίσως υπάρξουν δυσκολίες, διότι, ένα, διότι υπάρχουν μεγάλα προσκόμματα από τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στην τεχνολογία υγείας. Μπορούμε και να μην κάνουμε επικαλύψεις, αλλά να δούμε πώς ε, θα κάνουμε έρευνα, τι προτεραιότητες ε, θα δώσουμε στην έρευνα, τι επάρκειες υπάρχουν και βεβαίως να βελτιώσουμε και την ποιότητα της έρευνας. Ως προς ε, τη, τα, διάφορα medical devices, τις ιατρικές συσκευές, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ε, μία σωστή αξιολόγηση του τελικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, του ιατρικού προϊόντος. Πρόκειται για έναν αναδυόμενο τομέα και γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπε και ο κύριος Πέτερ Λίζε, υπάρχουν ίσως κίνδυνοι, αλλά θα πρέπει να δούμε, όπως είπε η κυρία Γκροστέτ, πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την ποιότητα υπέρ των ασθενών. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη συνένεση, διότι υπάρχει η επαρκής ευαισθητοποίηση για να επαγρυπνήσουμε υπέρ των ασθενών και να καλύψουμε τα συμφέροντα όλων των τομέων και όλων των ε, εμπλεκόμενων φορέων. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 13 Σεπτεμβρίου θα ε, ψηφίσουμε ε, στην ΕΜΒΗ, στην έκτακτη συνάντηση και μετά στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Άρα ολοκληρώνουμε με την ημερήσια διάταξη μέχρι τις 5 παρατέταρτο όπου προβλέπεται η ψηφοφορία για τις ανανεώσιμες. Θα σας δώσω μισή ώρα. Ε, αναστέλουμε τη συνεδρίαση μέχρι εκείνη την ώρα, 5 παρατέταρτο.

που Όχι, Hello everyone. You know we have only one vote. Ξέρετε ότι έχουμε μόνο μια ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Ερωτώ. Να γίνει ψηφοφορία. Είσαστε έτοιμοι. Ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, γι' αυτό χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας. Να ψηφίσουμε για την προσωρινή συμφωνία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδιατύπωση. Μία ψηφοφορία. Μία και μοναδική. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Και πέρας. Από την άλλη, από την άλλη. Την κάρτα σας. Θα σας μετρήσουμε, εν πάση κυρία Ελιόρ. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπας Έικαουτ. Και έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Τα λέμε στους συντονιστές αύριο το πρωί και μετά στις 10 ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Αύριο το απόγευμα έχουμε και τον Υπουργό της Αυστρίας. Παρακαλώ να προσέλθετε αθρώοι.